We start? Yes, okay. Monsieur le marteau Chers collègues, je déclare ouverte notre réunion conjointe. Κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ε, Προπολογισμού και ΕΚΟΝ τώρα, τώρα ξεκινάει. Θα πρέπει να αποφαθούμε ε, για το αποτέλεσμα των τεσσάρων τριμερών διαλόγων που έλαβαν υπόψη για το πρόγραμμα EU Invest. Θέλω να εξασφαλίσω ότι δεν έχετε παρατηρήσει για την ημερήσια διάταξη. Επίσης, θα πρέπει να αποφανθείτε για το σχέδιο πρακτικών της συνεδρίασης της 13ης Δεκεμβρίου, 29 ε, Ιανουαρίου και την συνεδρία του Φεβρουαρίου. Ε, εάν δεν έχετε παρατηρήσεις, εγκρίνονται τα πρακτικά. Τα μέλη της ομάδας που έπρεπε να αποφανθεί για το πρόγραμμα EISF θεωρούν ότι δεν μπορούν να αποφανθούν πριν από το τέλος ε, της ε, κοινοβουλευτικής θητείας. Η ΣΥΝ συγητέ του σχεδίου RSP, μετά από τις συνεδρίες των σκιωδών συνεδριάσεων και μετά από πολλές ημερείς συνεδριάσεις, θεωρούν ότι δεν υπάρχει πιθανή συμφωνία πριν την επόμενη συνεδρίαση και πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας. Η Επιτροπή ε, μοιάζει να ετοιμάζει μία συγχώνευση αυτών των δύο προγραμμάτων ή ένα είδος συγχώνευσης. Και επομένως τα μέλη, οι συνεισηγητές και οι σκιώδεις εισηγητές ε, εν τη σοφία τους αποφάσισαν ότι δεν θα πρέπει να κλείσουν το σημείο αυτό πριν το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας. Και τώρα θα πρέπει να αποφανθούμε πάνω στην έκθεση InvestEU και πάνω στις ε, διαθεσμικές διαπραγματεύσεις. Μετά από τέσσερις τριμερείς διαλόγους υπάρχει μερική συμφωνία για το InvestEU. Θέλω να συγχαρώ την ε, διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου. Να υπενθυμίσω ότι το Κοινοβούλιο περιμένει από το Συμβούλιο την επίσημη επιστολή που αναφέρει όλα τα common understandings, την, τα σημεία συνεννόησης για την, ε, τα τομιακά στοιχεία του CFP και ε, για το Investing You και με βάση τελευταίες πληροφορίες το Συμβούλιο συμφωνεί να δεχτεί τις πιστώσεις όπως προτείνει η διαπραγματευτική ομάδα. Αλλά δυστυχώς ε, επειδή είναι και πρωταπριλιά, <laughs> δεν ξέρω μήπως είναι αστείο τελικά, δικό αστείο. Και τώρα. Η Περβάνς στέλνει το λόγο. Ευχαριστώ. Μας ανακοινώσατε, Πρόεδρε, μια διαδικαστική πρόταση, ουσιαστικής φύσεως. Κατά τη διάρκεια δηλαδή αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας δεν θα αποφανθούμε για την, το θέμα της σταθεροποίησης, ούτε για το πρόγραμμα διαρθρωτικών αλλαγών που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια και είναι τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΟΝ και κυρίως η, η τελευταία κοινή συνεδρίαση ΕΚΟΝ και Μπουτς, νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε τους λόγους ε, που μας όθησαν σε αυτή την ε, εγκατάλειψη, σε αυτό το standstill. Καταρχάς θέλω να αποτίσω φορό τιμή στους συνεισηγητές. Ο Ράιμον Μπέγκε ήταν αρχικά και μαζί με αυτό ε, υποβάλαμε μια σημαντική πρόταση για να βελτιώσουμε την ταπεινή, κατά την άποψή μας, εισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τότε που πήρατε τη σκητάλη, από τις συζητήσεις μας προκύπτει ότι οι συνθήκες για να ενισχύσουμε αυτή την αρχική πρόταση της ε, Κομισιόν και να διατηρήσουμε την ιδέα της α, ε, λειτουργίας της σταθεροποίησης. Δεν, δεν μας την εγγυάται κανείς και καλό θα ήταν να αφήσουμε το φάκελο ως έχει. Λυπάμαι παρόλα αυτά για το γεγονός ότι οι εργασίες του Συμβουλίου γίνονται ε, αγνοώντας μας εντελώς. Και ο κίνδυνος είναι να φτάσουμε σε μια προσέγγιση ακόμα πιο διακυβερνητική, σε ένα τομέα όπου το έλλειμμα δημοκρατικότητας είναι ήδη πολύ ψηλό. Και γι' αυτό το να λάβουμε υπόψη, το να λάβει το Συμβούλιο υπόψη την άποψη του Κοινοβουλίου είναι εκ των όνων κάνευ. Αυτό σημαίνει ότι οι διάδοχοί μας θα πρέπει να εξασφαλίσουν αυτή τη λειτουργία της σταθεροποίησης. Να σας υπενθυμίσω, από ό,τι θυμάμαι, ότι την πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησε ότι το ευρώ χρειάζεται, από, χρειάζεται μια λειτουργία σταθεροποίησης ήταν το 1998. Σήμερα έχουμε φτάσει στο 2009, λέει η ομιλητρία, εννοεί 19 βέβαια, δεν υπάρχει ακόμα αυτή η λειτουργία. Και δεν θα ήθελα να ξυπνήσουμε κάποτε με επιζήμιες ε, συνθήκες για την Ευρωζώνη. Θα προτιμούσα λοιπόν να αφήσω την πρόταση πάνω στο τραπέζι ως έχει, μαζί με τις τροπολογίες που εκπονήσαμε με τον Ράιμουντ Μπέγκε, μαζί με τις συνεισφορές που ε, υπέβαλαν και οι άλλες ομάδες, παρά να σκοτώσουμε αυτή την ιδέα που πάντα υπήρχε σε αυτό το κοινοβούλιο. Να υπάρχει δηλαδή αυτή η λειτουργία της σταθεροποίησης. Ναι, υπήρχε μια βεβαιότητα, αλήθεια είναι, για την δυνατότητα θετικής ψήφου στην Ολομέλεια του Στρασβούργου σε δύο εβδομάδες. Και η πιθανή απόρριψη μιας τέτοιας πρότασης θα ήταν πραγματικό κρίμα, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, όπως τονίσατε κι εσείς. Σε ό,τι αφορά την ικανότητα να μας ακούει το Συμβούλιο, να μας λαμβάνει υπόψη, βλέπουμε πώς εκδηλώνεται σε όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτική θητείας. Ε, ούτως ή άλλως βλέπουμε τι άποψη, θα δούμε τι άποψη θα δώσει το Συμβούλιο για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και για τα τομεακά θέματα. Δεν θέλω να προδικάσω τα χειρότερα, αλλά διερωτώ με αν είναι έτοιμο το Κοινοβούλιο να ακούσει τα επιχειρήματα τα οποία υπενθυμίζουμε σε κάθε ε, συνεδρίαση του ΓΚΑΚ, του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Γιατί μπορεί να συνεδριάσουν κάποια στιγμή αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και να αποφασίσουν για το σύνολο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και για τα τομεακά προγράμματα. Γι' αυτό πρέπει να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ και πολύ προσεκτικά όλα αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως η θέση των ε, συνσηγητών είναι σωστή. Δηλαδή αυτή η λειτουργία, αν θέλετε, σταθεροποιητική, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντική κατά τη δική μου άποψη και αποτελεί έναν πολύ βασικό ε, πυλώνα για την εύρυθμη λειτουργία της ε, ε, ζώνης του ευρώ. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να διατηρηθεί αυτή η λειτουργία και θα πρέπει να αφήσουμε το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει τον απαραίτητο αγώνα έτσι ώστε να διασφαλίσει την ε, συνέχιση της μεταρρύθμισης ε, της ε, Ευρωζώνης, δηλαδή την δημιουργία των κατάλληλων εργαλείων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κρίσεων με καλύτερο τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Ας περάσουμε στις ψήφους τώρα. Στις καταρχήν, καταρχήν σε ό,τι αφορά το ΕΦΣΑΕΡ αλλά καταρχήν θα κάνουμε ένα τεστ, μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Άρχεται λοιπόν η δοκιμαστική ψηφοφορία. Πέρασε is closed. Σας ευχαριστώ. Περνάμε λοιπόν τώρα στην ψήφιση του αποτελέσματος της Σημερικής Συμφωνίας σε ό,τι αφορά το Invest EU. Και εδώ θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τον Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντε, τον συνεισηγητή μου και όλους τους σκιώδεις συζητητέ ε, για αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα Νομίζω πως το Κοινοβούλιο έπαιξε εδώ αποφασιστικό ρόλο στη βελτίωση του σχετικού κειμένου και τώρα λοιπόν για την επόμενη περίοδο, την επόμενη δημοσιονομική περίοδο έχουμε ένα κατάλληλο πρόγραμμα το οποίο βέβαια χρήζει τον απαραίτητων ε, κονδυλίων, τη απαραίτητη πρικοδότηση από τον προπολογισμό. Πράγμα για το οποίο θα αγωνιστούμε από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Πάντω, ό,τι αφορά το περιεχόμενο, νομίζω πω επιτύχαμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και γι' αυτό σα ευχαριστώ ευχαριστώ όλου για τη συνεισφορά σα, ε, για την ε, θετική έκβαση λοιπόν των διαπραγματεύσεων. Άρχεται η ψηφοφορία ονομαστικά. Πέραση 40 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν. Συγχαρητήρια σε όλους μας. Ευχαριστώ. Very good. Πολύ ωραία. Ήταν ε, πολύ σύντομη λοιπόν αυτή η κοινή συνεδρίαση Επιτροπών Έκων και Μπάτζ. Σύντομη αλλά πολύ ενδιαφέρουσα. Ε, και ε, λίγα, ε, μια στιγμή δώστε μας απλά για να αποχωρήσουν οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Μπούτζη, από την αίθουσα, ώστε να συνεχίσουμε με τις εργασίες της